εκ μέρου τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά πώ είναι δυνατόν με τόσο κόσμο που έχετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην βρήκε κανεί το χρόνο μια τόσο σημαντική μέρα σαν τη σημερινή να έρθει εδώ στην Υποπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εσεί όμω παραμείνατε εδώ όλο το πρωί και έτσι ευχαρίστω σα δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, είμαστε εδώ και παραμείναμε εδώ γιατί είναι θέματα τα οποία μα ενδιαφέρουν. Είμαστε και εμεί σε διαδικασία μεταρρύθμιση η πρώτη προφορική ερώτηση που απαντήθηκε είναι σχετική. Τα ανθρώπινα δικαιώματα εμείς τα βάζουμε σαν προϋπόθεση. Ε, δεν ε, κάνουμε εξαγωγές εφόσον δεν τηρούνται αυτά. Θέλω να απαντήσω στην κυρία Λοχμπίλερ όμως. Η έλεγχη εξαγωγών αποτελεί ένα μέσο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αν γνωρίζουμε ότι ένα κράτος δεν έχει τις προδιαγραφές που απαιτούνται για τη χρήση της τεχνολογίας, έχουμε και άλλα μέσα. Έχουμε τις κυρώσεις, άρθρο 15 της συνθήκης, και μπορούμε επίσης να κοιτάξουμε και το ευρύτερο πλαίσιο των εργαλείων που έχει διαθεσή της Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, για τη γενική μας διεύθυνση, πρέπει να ξέρετε ότι βεβαίως και θέλουμε να είμαστε εδώ και να παρακολουθούμε τις συζητήσεις σας που είναι τόσο ενδιαφέρουσες. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Έχουμε ήδη μαζί μας τον επόμενο προσκεκλημένο μας για να συζητήσουμε για τη Βόρεια Κορέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, όλους τους προσκεκλημένους για τις εξαίρετες παρουσιάσεις σας, παρόλο που είχατε λίγο χρόνο στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ.